μια προφορική ερώτηση. Τι είναι το κοινωνικό τριπλό αλφα στον κοινωνικό τομέα. Και δίνω το λόγο στον συντάκτη της ερωτήσεως, κύριο Χέντελ, πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη χρειάζεται κατεπηγόντως ένα κοινωνικό τριπλό α. Αναμφίβολο αυτό. Και άλλωστε το έχει και η Επιτροπή αποδεχτεί. Οι πάτες γνωρίζουν ότι η ψηλή ανεργία μπορεί να θεωρείται ανώδυνη αν μειώνεται ελαφρά και καταγράφεται αυτό ε, στα επίσημα στατιστικά στοιχεία αλλά λησμονούμε ότι ε, με την υποβάθμιση της κοινωνικής προστασίας έχει φτάσει το όριο της φτώχειας σε επίπεδα απαράδεκτα και για τον όσα και οι νέοι ε, πολύ δύσκολα μπορούν να φτάσουν σε μια θέση εργασίας και αν βρουν θέση εργασίας είναι από αυτές τις προσωρινής απασχόλησης που εργάζεται κανείς σε συνθήκες φτώχειας. Φαίνεται ότι η Επιτροπή είναι σε θέση τώρα να αντιληφθεί και να αναλάβει μια πρωτοβουλία για το κοινωνικό τριπλό τον Οκτώβριο του 2014 ο Ζων Κλώτ Ιουνκέρ είχε περιγράψει φιλόδοξα σχέδια εν προκειμένου. Και μέσα στην έκθεση των πέντε προέδρων επίσης για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απασχόληση και τα κοινωνικά. Το 2015 έχουμε την περιγραφή του οράματος ενός ευρωπαϊκού τριπλού κοινωνικού αλφα και, περιγρα... και περιγράφεται ως εξή ε, να αξιοποιηθεί το μέγιστο δυναμικό για να αντιμετωπιστούν μεγάλες κοινωνικές ε, προκλήσεις και προκλήσεις για την απασχόληση με κοινέου στόχους, κοινωνικούς στόχους απασχόλησης στην Ευρώπη, στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Λόγια. Όλα αυτά είναι λόγια. Και η Επιτροπή νομίζω ακόμα δεν συζητά καν τα κοινωνικά ζητήματα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν απλές λύσεις, δεν υπάρχουν γενικές λύσεις για τα κοινωνικά ζητήματα στην Ευρώπη. Αλλά και στην πρώτη ακόμη ε, την πρώτη αυτή προεξαγγελία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν την έχει υλοποιήσει. Δεν υπάρχει καν ενημέρωση διαρθρωμένη για το κοινωνικό τριπλό Α. Και τώρα έχουμε μια ανακοίνωση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΜΕΝ, αλλά κυρία Επίτροπε, κυρία Τάισεν Αυτή η σημερινή διαρθρωμένη ενημέρωση δεν νομίζω ότι μας φώτισε. Εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω να υπάρχει ενημέρωση για σαφή πρόθεση του τι θα συμβεί από εδώ και μπρο. Μπορεί γενικόλογα και κοινόλογα πράγματα να ακούσαμε. Ωραία έχεις για τα αυτιά όλων μας. Αλλά πείτε μας τι είναι το κοινωνικό τριπλό αλφα. Ποιε είναι οι συγκεκριμένε λεπτομέρειε για την έννοια, τα συστατικά της, τους στόχους της. Τρίτον, ποιοι είναι οι φυστάμενοι και κυρίως ποιοι είναι οι νέοι μηχανισμοί. Οι διαδικασίες, οι δείκτες, τα μετρήσιμα βήματα εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την υλοποίηση των στόχων. Τέταρτον, πώς θα υλοποιηθούν τα μέσα. Πέμπτον, ποιο είναι το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για το κοινωνικό τριπλό. Α, έκτον, ποια θα είναι η καλύτερη κοινωνική σύγκληση προς τα άνω επί τη βάση κοινών προδιαγραφών υψηλού επίπεδου που πρέπει να προωθούν. Όλα αυτά είναι οι ερωτήσεις που έχουμε διατυπώσει και στην Επιτροπή μου, αλλά υπάρχουν και άλλες τι μεταρρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα προαγάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια καλύτερη κοινωνική σύγκληση. Έκτον, όγδον, συγγνώμη. Ποιες είναι οι πρόοδοι, ε, ποιος είναι ο τρόπο με τον οποίο θα επαληθεύονται αυτέ οι πρόοδοι. Και εν τέλει, πώς θα σχεδιάσει και θα εγκαθιδρύσει ένα κοινωνικό τριπλό αλφα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο για την ε, Ευρωζώνη. Δεν θέλουμε δηλαδή μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Αυτέ είναι οι μεγάλε προκλήσεις, αυτά είναι τα μεγάλα ερωτηματικά και πιστεύω ότι η κοινωνική κατάσταση είναι το κέριο εκείνο ερώτημα, το καθοριστική σημασία σε εκείνο ερώτημα που θα κρίνει την επιβίωση μιας κοινωνικής και αλληλέγγυας Ευρώπης. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε στο Μάρτιο του 2017. Δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε να εκδοθεί λευκή βίβλος. Τώρα χρειάζονται συγκεκριμένα, απτά, σαφή βήματα για να προχωρήσουμε προς μια κοινωνική Ευρώπη. Και ευχαριστώ για την προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στην Επιτροπή, βασικός μας στόχος είναι μια Ευρώπη με τρία αλφα σε επίπεδο κοινωνικό. Είναι πραγματικά όχι μόνο στόχος, όχι μόνο φιλοδοξία, αλλά υποχρέωση η οικονομική μας ανάπτυξη να συμβαδίζει με τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Αυτός είναι ο πυρήνας του κοινωνικού μας προτύπου και της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Ένα τριπλό κοινωνικό αλφα απαιτεί να υπάρξει μια πορεία ισορροπημένη με στόχο την δημιουργία σωστών θέσεων απασχόλησης και προστασία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασιακής του ζωής. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές συνέπειες σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής. Μόνο τότε θα πετύχουμε την κοινωνική Ευρώπη. Λάβαμε ήδη τα πρώτα μέτρα έτσι ώστε να οδεύσουμε προς την συγκεκριμένη αυτή κατεύθυνση. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο συμπεριλαμβάνουμε την ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών επιδόσεων Κάνουμε επίσης μελέτες επιπτώσεων σε κοινωνικό επίπεδο και στα πλαίσια του προγράμματος για την Ελλάδα κάνουμε συστάσεις προς τα διάφορα κράτη-μέλη και την, για την επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας. Προτείναμε και το Συμβούλιο δέχτηκε να αυξήσουμε την προχρηματοδότηση από το 1% στο 31% του Ταμείου για την Νεότητα, συνολικά μέχρι ένα δις. Και αυτό επέτρεψε το πρόγραμμα αυτό για την απασχόληση των νέων να ξεκινήσει με σωστούς τρόπους για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Θα υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες κατά τη διάρκεια της ε, ε, ε, εργασιακής τους δραστηριότητας. Επίσης και η νέα πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας θα συνεισφέρει στην βελτίωση των συνθήκων εργασίας των εργαζομένων οι νέες ρυθμίσεις θα βοηθήσουν επίσης αυτούς οι οποίοι αναζητούν θέσεις απασχόλησης να κινηθούν με μεγαλύτερη ευκολία. Και υπάρχει και σήμερα όπως ξέρετε το συζητήσατε νωρίτερα μια νέα πρόταση για την οδηγία σχετικά με τις αποσπάσεις των εργαζομένων. Ε, καλύτερη επίσης ε, ισορροπία ανάμεσα στις δυνατότητες ε, που υπάρχουν για γυναίκες και άνδρες και μια πιο συνολική αξιολόγηση των ισχυουσών οδηγιών έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω συνέργειες πριν από το καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε άλλωστε σήμερα μια μεγάλη διαβούλευση και για την Ευρωπαϊκή Χάρτα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος ο Ιούνκερ στο Σεπτέμβριο το είχε ανακοινώσει αυτό στην επίσημη ομιλία του. Ε, στην διαβούλευση θα συμπεριληφθούν και τα Εθνικά Κοινοβούλια και φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ζητώ όλους να πάρετε μέρος στη συζήτηση και να ε, εκφέρετε και εσείς τη δική σας πρόταση. Ζητούμε επίσης και από την κοινωνία των πολιτών. Θέλουμε να ενισχύσουμε τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Είμαστε, θυμίζω, η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και οι περισσότεροι από τους πολίτες έχουν υψηλά επίπεδα ε, προστασίας Πρέπει λοιπόν τα κοινωνικά δικαιώματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο να εφαρμοστούν πλήρως. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει είναι πάντα επίκαιρο και χρήσιμο. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά από την οικονομική κρίση και νομίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη στα κοινωνικά θέματα θα έλεγα θα παραμείνουν η αναφορά και στον 21ο αιώνα. Έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωζώνη, απαιτείται περαιτέρω σύγκληση και στα κοινωνικά θέματα και στα θέματα της αγοράς εργασίας είναι απαραίτητο για την αύξηση της αντοχής και της επίδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν κεντρικός στόχος για τις χώρες της Ευρωζώνης αλλά και οι υπόλοιπες χώρες μέλη φυσικά είναι προσκεκλημένες να συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, είμαι σίγουρη ότι αυτή η τακτική θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε στην απόκτηση του λεγόμενου τριπλού κοινωνικού αλφα. Ε, αυτό θα έχει συγκεκριμένες συνέπειες και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Έχουμε ήδη ξεκινήσει πάνω από 10 πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αναπτυχθεί τον 21ο αιώνα ακόμα περισσότερο το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο και να συνεχίσει να είναι χρήσιμο για τους Ευρωπαίους πολίτες και να συμβάλλει στην ανάπτυξη Νομίζω ότι υπολογίζουμε στην υποστήριξή σας και στη συνεργασία σας. μισή λεπτό κύριο Κάζα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Η πρόταση του τριπλού αλφα μπορεί να είναι μια συμβολή στην ευημερία των πολιτών και προφανώς μπορεί να εξελιχθεί Βάσει της συνθήκης, μεταξύ άλλων η Ένωση έχει το δικαίωμα να συμπληρώνει και να επικουρεί τα κράτη-μέλη σε τομείς όπως η υγεία, οι συνθήκες εργασίας, κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία. Ωστόσο, για να επιτευχθεί το εγχείρημα αυτό χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών με σαφείς στόχους και ορισμούς είναι χρήσιμο να θυμόμαστε ότι για την ομοιογενή ανάπτυξη χρειάζεται και την ε, κοινωνική συνοχή χρειάζεται ενωσιακή συνεργασία. Προφανώς πιστεύω και συμφωνώ ότι οι κοινωνικές παράμετροι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική δράση. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν στην κρίση που διανύουμε. Θέτοντας τους πολίτες σε κίνδυνο. Η προστασία των πολιτών μας είναι καθήκον. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή για τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν τους κοινωνικούς δείκτες στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης της Ένωσης για τα κοινωνικά θέματα και να χρησιμοποιεί τους δείκτες αυτούς ως μηχανισμό για να αναλάβει δράση. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για 1,5 λεπτό κυρία Στάινμπρουκ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του κύριου Γιούγκε, είχαμε μεγάλες προσδοκίες κυρία Τάισεν και μέχρι τώρα θεωρούμε ότι έχουν γίνει πολύ λίγα. Λίγο περισσότερο κοινωνικός χαρακτήρας, ε, κοινωνικός χαρακτήρας, κάποιες εκθέσεις ενδεχομένως και μια μη δεσμευτική δήλωση για την καταπολέμηση της ανεργίας. Τώρα μετά από ένα μισή χρόνο μπορούμε να πούμε ότι κάποιες πρωτοβουλίες υπήρχαν, αλλά με την αρχική αναγγελία που είχατε κάνει, λίγα συγκεκριμένα πράγματα έχουν γίνει για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα δώσουμε ένα κοινωνικό τριπλό α που θα έχει σχέση με αυτά που προσδοκούν οι πολίτες της Ευρώπης. Δεν βοηθάμε τους εργαζομένους με αυτά τα οποία κάνουμε στην αγορά εργασίας επικρατεί όλο και μεγαλύτερο κοινωνικό dumping. Θα πρέπει η Επιτροπή να καταπολεμήσει την επισφαλή εργασία, την ανεργία. Θα πρέπει να προσπαθήσει να αγωνιστεί κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Χρειαζόμαστε ένα ελάχιστο εισόδημα, μισθούς που θα επιτρέπουν μια αξιοπρεπή διαβίωση και θα πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη σημασία στον κοινωνικό διάλογο. Κατά πολέμηση της φτώχειας θα πρέπει να είναι βασικός σας στόχος για να μπορέσετε να δώσετε κοινωνικό τριπλό α στην Ευρώπη και στην αναθεώρηση της οδηγίας για τις αποσπάσεις και για το συντονισμό των κοινωνικών συστημάτων θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Γκέι και ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε στις τράπεζες δίνουμε τριπλό α για την σωστή οικονομική κατάσταση και ε, τα πιστοληπτικά ε, ε, ιδρύματα δίνουν αυτό το τριπλό α το οποίο εμείς τώρα δίνουμε στον κοινωνικό τομέα και χαιρετίζουμε αυτή την απόδοση της ένδειξης τριπλού κοινωνικού αλφα. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια έννοια για ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό όμως που δίνουμε στα λόγια θα πρέπει να ακολουθείτε και από έργα για να μην παραμένουν κενό γράμμα αυτά τα οποία δηλώνουμε. Θα πρέπει να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση. Πώς μπορεί να δοθεί ένα κοινωνικό τριπλό αλφα στην Ευρώπη. Τι ακριβώς πρέπει να συμπεριλαμβάνει. Τι πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη για να τα καταφέρει. Είμαι ανοιχτό σε μια τέτοια συζήτηση και θα ήθελα να κάνουμε περισσότερα από ό,τι μέχρι τώρα για να εμπλέξουμε και του πολίτε γιατί τα ε, ε, ε, συντηρητικά κόμματα στη Γαλλία ζητούν ε, ε, ε, ακριβώς αυτή τη διάσταση. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κ. Καλβετσέμπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την Επίτροπο. Καλησπέρα, Επίτροπε, καταρχάς. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι όταν η Επιτροπή χρησιμοποιεί λέξεις και ορολογία θα πρέπει να έχει σαφώς υπόψη τη πόσο σοβαρά είναι τα θέματα που θα αντιμετωπίσει. Ήταν λοιπόν πολύ αναγκαίο να ορίσει η Επιτροπή με πολύ σαφή τρόπο, τρόπο τι εννοούσε με το τρίπλο α, απλά και όχι να το χρησιμοποιεί απλά σαν μια λέξη, μια, ένα σύμβολο. Θα πρέπει λοιπόν να οριστεί η βούληση που έχουν. Ελπίζω, ελπίζω να μείνει αυτό σε ένα σύμβολο μιας πραγματικής βούλησης να δημιουργήσουμε μια κοινωνική Ευρώπη. Και ελπίζω η Επιτροπή να μην πέσει στην ιδέα να αρχίσει να ε, ανεβοκατεβάζει το τριπλό α στο 2 μείον, 2 συν 2 με μία κλίμακα. Και εν τέλει ποιος είναι ποια υπηρεσία, ποια εταιρεία είναι αυτή που θα δώσει τον αριθμό. Θα ήθελα να δώσει προτεραιότητα στον δρόμο για μια καλύτερη κοινωνική Ευρώπη. Θα σας καλούσα να μην μιλήσουμε μόνο για την απασχόληση, Ωστόσο, το πρώτο στοιχείο του τριπλού Α είναι η πλήρη απασχόληση. Α μιλήσουμε όμω για τι κοινωνικέ πολιτικέ. Μιλήστε για τη φτώχεια και τον τρόπο καταπολέμησή τη. Σήμερα, όχι αύριο. Μιλήστε για την κυκλοφορία των φοιτητών στην εκπαίδευση, Erasmus Plus κτλ. Σήμερα. Και παρακαλώ μην ξεχνάτε ότι η προστασία του εργαζομένου δεν σημαίνει προστατευτισμό. Κάποιο, κάποια τελευταία πρόταση. Τι αξιοπιστία θα έχει η Επιτροπή υποστηρίζοντας μια καλύτερη κοινωνική Ευρώπη με τριπλή, τριπλό α όταν με το κείμενο του κυρίου Τούσκ ε, για τη Βρετανία καταψηφίζει και αρνείται την ελεύθερη κυκλοφορία. Η κυρία Ζήμερ, ένα λεπτό, ένα μισή λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. στη Γερμανία και σε άλλα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια είχαμε θετική οικονομική ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά δεν άλλαξε η γενική εικόνα σε αυτές τις χώρες. Υπήρχαν ελλείμματα και αυτό δίνει ε, ε, ξεκάθαρα να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ε, κοινωνικής κατάστασης των πολιτών. Γι' αυτό το κύριο καθήκον για μας θα πρέπει να παραμείνει όπως είναι και μέχρι τώρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς συγκεκριμένα ως Ευρωπαϊκή Ένωση για τα 130 ε, εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν ε, σε όρια φτώχειας δεν θα πρέπει να μιλήσουμε μόνο για την αγορά εργασίας. Θα πρέπει ευρύτερα να δηλώσουμε ποια είναι τα συγκεκριμένα κριτήρια που θέλουμε, γιατί θέλουμε μετρήσιμα κριτήρια για την καταπολέμηση της φτώχειας δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για δημιουργία θέσεων απασχόλησης χωρίς να το συνδέουμε και με ένα ελάχιστο μισθό που θα οδηγεί στην καταπολέμηση της φτώχειας. Θέλουμε συντάξεις που να καταπολεμούν τη φτώχεια, διαφορετικά δεν έχει νόημα. Θα πρέπει να δούμε αυτή την ισορροπία μεταξύ της ευελιξίας και της ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια αυτή η flexicurity οδήγησε σε μεγαλύτερη φτώχεια και σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να εξετάσουμε για να καταπολεμήσουμε την φτώχεια. Δεν θα πρέπει να μιλάμε για ελάχιστα δικαιώματα, αλλά για βασικά θεμελιώδη δικαιώματα. Κάθε άνθρωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα σε κοινωνική ζωή χωρίς φτώχεια. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να σας κόβω, αλλά έχουμε περιορισμούς στο χρόνο. Παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο σας. μιση λεπτό. Η κύριε Λαμπέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε. Όταν ξεκινήσαμε να συζητούμε για κοινωνικό τυπλό α, κάποιοι άρχισαν να ήλπιζαν πέρσι ότι θα υπήρχε κάτι καλύτερο για την κοινωνική Ευρώπη. Και θα στηριζόταν περισσότερο στη δουλειά που είχαμε κάνει στο παρελθόν για θέματα που δεν ήταν μόνο το ΑΕΠ. Γιατί εδώ αντλούμε από το πώς ε, βλέπουμε το θέμα του τριπλού α. Η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης χτυπήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια και το κοινοβούλιο ήταν σαφές. Το θυμάστε κι εσείς, κύριε Επίτροπε. Ήταν αποδεκτό γενικότερα ότι οι πολλές περικοπές οδηγούν σε, σε ξέραμα του φυτού που θέλουμε να μεγαλώσουμε. Εμείς που έχουμε την εμπειρία της φτώχειας μπορώ να σας πω ότι δεν έχει γίνει επαρκής διαβούλευση και ένα βασικό θέμα είναι η αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Στην αγορά εργασίας βλέπουμε να μειώνονται οι θέσεις, μειώνονται οι ευκαιρίες δουλειάς και αντιμετωπίζω μια σειρά προκλήσεων. Ελπίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη θα προχωρήσουν επικοδομητικά στον τομέα αυτό. Αυτό το θεωρούν δεδομένο οι Βρετανοί. Ωστόσο υπάρχει ένα θέμα υλοποίηση σε ό,τι αφορά τη μελλοντική ε, νομοθετική δράση. Αφορά όλη την Ευρώπη ή το κέντρο της Ευρώπης. Μιλούμε για μια σειρά εξαιρέσεων στη Βρετανία για την ε, οδηγία για την ε, παιδική μέρημνα, για την οικογενειακή μέρημνα. Αυτό είναι δύο, Ευρώπη δύο ταχυντήτων. Η κυρία Ατζέρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λυπάμαι κύριε Επίτροπε, δεν συμφωνούμε. Ήμουν πεπισμένη ότι αυτό που ήταν μια ένδειξη και μια κουβέντα του Πρόεδρου Γιούνκερ όταν είχε έρθει εδώ δεν είχε καμία υλοποίηση. Μιλάτε για ένα τριπλό κοινωνικό α, σαν ετικέτα. Σαν αυτό να χρειάζεται μια Ευρώπη που πεινάει, που βρίσκεται στα όρια των δυνάμεών της και όπου όχι πια η φτώχεια αλλά η αθλειότητα αποτελούν συνθήκη ζωών, ζωής εκατομμυρίων πολιτών. Δεν μπορούμε να μιλούμε για τριπλή, τετραπλή, πενταπλή α αν δεν μιλήσουμε, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για προβλήματα, για συγκεκριμένες λύσεις ε, που χρειάζονται οι οικογένειες που πεινάνε. Λέτε, γίνανε προτάσεις. Ξέρετε ποια είναι η τελευταία. Ότι σήμερα η Επιτροπή ζήτησε αλλαγή του προπολογισμού του 2016 της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Φιλανδίας, της Ρουμανίας και του Βελγίου. Για ποιο λόγο? για σοβαρές παρεκκλήσεις από τους στόχους λιτότητας που έχουν συμφωνηθεί. Αυτό είναι το τριπλό α που επιβάλλεται και άλλες διαθροτικές μεταρρυθμίσεις, περικοπές και σας θυμίζω ότι δεν είναι αυτά τα μέτρα που εξασφαλίζουν την επιβίωση, την ύπαρξη εκατομμυρίων πολιτών που πεινούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Μαρτά. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Τσίμερ, το να βάλετε το κοινωνικό κομμάτι στο ίδιο επίπεδο με το οικονομικό είναι το καινούριο σύμβολο που κοροϊδεύει όμως ο κύριος Γιούνκερ. Οι πολίτες γίνονται όλο και πιο ευρωσκεπτικιστές. Αυτή η αλλαγή θέλει να αναπτύξει και το κράτος πρόνοια σύμφωνα με δύο άξονες, διασφαλίζοντας την κοινωνική προστασία αλλά προσπαθώντας ε, να καθορίσουμε και κοινού στόχους για την κοινωνική σύγκληση στο σύνολο της ζώνης ευρώ. Αν αυτό το πρότυπο του να προσδέσει κανείς κάτι το κοινωνικό σε ε, μια συνάντηση κορυφής επιτρέψει να γίνουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, βασικός στόχος παραμένει πάντα η οικονομική σύγκληση στη ζώνη ευρώ που ε, φαίνεται ότι αντιμετωπίζει με πολύ σκεπτικισμό την κοινωνική Ευρώπη. Ε, η βελτίωση των κοινωνικών συνθήκων φαίνεται ότι θα θέσει σε κίνδυνο την ισορροπία της αγοράς εργασίας, κάτι το οποίο θα είναι δύσκολο να συνδυαστεί με πολιτικές για μια αγορά εργασίας πιο αποτελεσματική σε μια εποχή δραστικών δημοσιονομικών πιέσεων που επαναλαμβάνονται συνεχώς από το 2007 και δημιουργούν μια ενδημική φτώχεια. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Ζαριανόπουλος. Με τριπλό αλφα ή και αξιολόγησης αξιολογούν κερδοφόρες τράπεζες, οικονομίες, επενδύσεις. Με το κοινωνικό τριπλό α, δηλαδή δίθεν κοινωνικά κριτήρια στο σφαγείο των εργατικών δικαιωμάτων που λέγεται Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοροϊδεύει και προκαλεί. Αλλά ομολογεί κιόλα ότι η φθηνή ευέλικτη εργασία είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το κεφάλαιο. Ούτε ευχολόγια, ούτε δίθεν δημοκρατική λογοδοσία σε αντιδραστικά όργανα όπως το Ευρωκοινοβούλιο εξανθρωπίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράδειγμα, ακούστε ορισμένε απαντήσει τη Επιτροπή σε ερωτήσει του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, δεν καθορίζει δικαίωμα σε μόνιμε συμβάσει εργασία, δηλαδή δουλειά λάστιχο για ψίχουλα. Άλλοι, σε προγράμματα του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν μισθό ούτε βέβαια ασφάλιση. τζάμπα και ανασφάλιστη εργασία ενώ το σύστημα eures υπονομεύει τη μόνιμη εργασία ενισχύοντας τα δουλεμπορικά γραφεία. παράδειγμα η ελλάδα όπου με την αξιολόγηση του τρίτου μνημονίου κυβέρνηση και κοαρτέτο παραπλανώντας για ευρωπαϊκή ένωση πιο φιλολαϊκή από το διεθνές νομισματικό ταμείο για ενδιαφέρον για τους πιο αδύναμους μοιράζουν φτώχεια ανάμεσα σε και πετσοκόβουν πάλι μισθούς συντάξεις κοινωνικά επιδόματα και δαπάνες βάζουν τα φόμπλακα στην κοινωνική ασφάλιση και τα εργασιακά δικαιώματα. καμιά απορία εδώ στελέχη της ένωσης και όλων των κυβερνήσεων ξεδιάντροπα καλούν για αξιοποίηση της πάνθηνης δουλειάς των προσφύγων αν ξεφύγουν από τους βομβαρδισμούς τους πνιγμούς τα hot spot την απέλαση και τον εγκλωβισμό στην ελλάδα. ο μονόδρομος για τους λαούς είναι η απαλλαγή από αυτή την πολιτική και από την εξουσία του κεφαλαίου. κυρία Μόρα Σότιε, ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρία Επίτροπε, το 2014 όταν είχε η Κομισιόν να μας αναγγείλει στο Κοινοβούλιο την ωραία αυτή έκφραση και τη βούλησή της να δημιουργήσει την κοινωνική Ευρώπη με ένα τριπλό α, είχε αποτελέσει τεράστια ελπίδα για μας αλλά και για το λαό της Ευρώπης. Ο δικός χάρτης που είχατε διαμορφώσει πριν λίγο μας ε, δείχνει να καταλάβουμε πόσο δουλεύετε για το στόχο αυτό καθημερινά. Τα στοιχεία έχουν μικρά βελτίωση, αλλά έχουμε πάντα 9% ανέργων στην Ευρώπη κατά μέσο όρο, πολύ περισσότερο από ό,τι στις είπα. Η ανεργία των νέων φτάνει τα 20%, ανησυχητικό, πολύ περισσότερο σε κάποιες χώρες 25% των πολιτών μας ε, κινδυνεύουν πάντα να πέσουν στο επίπεδο της φτώχειας. Η κοινωνική Ευρώπη περνά προφανώς από την επαγγελματική ένταξη. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας πω ότι το πρώτο εργαλείο της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής Ευρώπης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων, η εγγύηση νέων, Ελπίζω ότι όλα μαζί στο πρόγραμμα που περιγράψατε θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να διατηρήσουμε τα εργαλεία αυτά. Πρέπει να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη, διότι τα κράτη είναι αυτά που καθυστερούν στην οικοδόμηση από κοινού της κοινωνικής Ευρώπης, που είναι και η Ευρώπη της απασχόλησης και η Ευρώπη της κοινωνικής προστασίας όλων των πολιτών. Ευχαριστώ που δουλεύετε το θέμα αυτό και να υπολογίσετε σε εμάς. Η κυρία Ούλσοκ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Και ευχαριστώ την Επιτροπή για την πρωτοβουλία σας. Προφανώς θα απαιτήσει πολλά από μας αν θέλουμε να πετύχουμε αυτό το τριπλό κοινωνικό αλφα. Ποιοι είναι, ποιοι είναι οι όροι, ποιε είναι οι προποθέσει ενό τριπλού Α σε μια περίοδο μεταναστευτική κρίση, υψηλή ανεργία, περικοπή περιορισμών των μέσων ενημέρωση και μια οικονομική κρίση που δεν έχει προχωρήσει. Ταυτόχρονα οι κοινωνικοί εταίροι δεν εμπλέκονται όπως θα όφυλαν και θα έπρεπε για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο χωρίς αυτό μόνο στην πολιτική. Και πιστεύω ότι οι, πρόσφατες, οι εμπειρίες των πρόσφατων ετών είναι παράδειγμα. Η Ευρώπη έχει κάνει σημαντική δουλειά, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται στις χώρες που αντιμετώπισαν κρίση που διοικούνται από την Τρόικα και υποχρεώθηκαν να απομακρυνθούν από τα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Οι χώρε αυτέ είναι σε χειρότερη κατάσταση τώρα από άλλε, γιατί οι κοινωνικοί εταίροι δεν μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους. Πρέπει να επιτρέψουμε λοιπόν στους ανθρώπους να συνεργάζονται, να δουλεύουν ελεύθερα με πολιτικούς, με συνδικάτα για να αποκαταστήσουμε το παλιό σύστημα. Η κυρία Λόπε Φοντανιά, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε. Πέρασαν πολλοί μήνες από τότε που ο πρόεδρος Γιούνκερ μίλησε για πρώτη φορά για το τριπλό κοινωνικό α. Είναι σαφές ότι όταν το ανήγγειλε θεωρήσαμε ότι η ιδέα ήταν πολύ καλή. Η πλειοψηφία των βουλευτών ωστόσο δεν κατάλαβαν επαρκώς ποια θα ήταν η πορεία που θα ακολουθούσε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σαφείς έννοιες αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Οι Ευρωπαίοι πολίτες χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν και να υποστούν πολλές θυσίε κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η βελτίωση της κρίσης, η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και η ανάπτυξη θα πρέπει να περάσει στην κοινωνία, ιδίω στα άτομα που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Αν το τριπλό α σημαίνει ότι η Ένωση μέσω των κρατών μελών θα δουλέψει για μια μεγαλύτερη κοινωνική σύγκληση, περισσότερες θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι ευπρόσδεκτη. Για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο περιλαμβάνει ένα σύνολο κοινωνικών δικτών που αναδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία για κοινωνικά θέματα. Ωστόσο, για να πετύχουμε την, τα χαρακτηριστικά αυτά χρειαζόμαστε σαφείς δείκτες που μπορούν να αναλύσουν σωστά την πρόοδο που επιτεύχθηκε και κυρίως να προσανατολίζουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές προς, την, το τριπλό α, όταν είμαστε ακόμα μακριά από την στρατηγική του 2020. Ευχαριστώ την Επιτροπή και την Επίτροπο κύριο Τίσεν για τις εξηγήσεις της και ελπίζω η πρωτοβουλία αυτή να πετύχει. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό η κυρία Γιουγκέριος. Ευχαριστώ πολύ. Έχω τρεις ερωτήσεις. Ποια είναι αυτή η ευρωπαϊκή αγορά απασχόλησης όταν πρέπει κανείς να δουλεύει σε δύο δουλειέ για να πληρώσει του λογαριασμού του. Όταν δεν καταφέρνουμε να βρούμε δουλειά, τι νόημα έχουν όλα τα υπόλοιπα και τα ελάχιστα που μπορεί να κερδίζει κανείς σε ένα εργοστάσιο ειδών ρουχισμού στην Ευρώπη δεν ανταποκρίνονται σε μια κοινωνική Ευρώπη. Θα πρέπει η αγορά εργασίας να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες μας για μια Ευρώπη που θα τους περικλείει όλους. Να μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε πάντοτε νέοι και καλά στην υγεία μας. Πρέπει να μιλάμε για την καταπολέμηση της φτώχειας και θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων, να ισχύουν συλλογικές συμβάσεις, να τηρούνται και να μην έχουμε μια πολιτική à Θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν, κυρία Επίτροπε, να αναλάβετε δράση. Ο κύριος Όγκορ, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτως με την φιλοδοξία της Επιτροπής να έχει και κοινωνικά μέτρα που θα συνοδεύουν τις μακροοικονομικές πολιτικές και καταλαβαίνω και υποστηρίζω το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική πρόοδος συνδέονται και αλληλοενισχύονται. Όταν μιλάμε για τον ορισμό του κοινωνικού τριπλού Α, συμφωνώ επίσης απολύτω με την ιδέα μιας οικονομικά ισχυρής Ευρώπης που θα έχει οικονομική ανάπτυξη, που θα παρέχει θέσεις απασχόλησης και θα βελτιώνει τη ζωή των πολιτών. Παράλληλα, κατά την προσπάθειά μας να επιτύχουμε αυτό το στόχο θα πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική νομοθεσία, την υπερβολική ρύθμιση που θα μας αποτρέπει από το στόχο μας και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη, την ανάγκη προστασίας της ελεύθερης αγοράς και την διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό. Ο κύριος Πυρίνσκι. Thank ε, ε, Επίτροπε, νομίζω ότι θα πρέπει να θυμηθούμε τι είχε πει ο κύριος Γιούνκερ, ο πρόεδρος Γιούνκερ τον Οκτώβριο του 2014. Θέλω η Ευρώπη να αφιερωθεί στο να είναι σε κοινωνικό επίπεδο, όπως επίσης είναι στον τομέα της οικονομίας. Η ερώτησή μου, Επίτροπε, είναι η εξής. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την προσπάθεια αυτή στα κοινωνικά θέματα σε σχέση με τα μακροοικονομικά και χρηματοπιστωτικά. Στην ομιλία σας στο Λουξεμβούργο τον προηγούμενο Ιούνιο, στην ερώτηση υπάρχει μια νέα κοινωνική Ευρώπη, είπατε ένα πανηγυρικό ναι. Δυστυχώς όμως εγώ νιώθω ότι η πραγματική απάντηση είναι ένα εξίσου αποφασιστικό όχι. Η πραγματική προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως περιλαμβάνεται ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ε, η λιτότητα, συνεχής πίεση έτσι ώστε να προχωρήσουμε στις λεγόμενες διαφθρωτικές και δημοσιονομικές ισορροπίες και οι κοινωνικές πλευρές και οι συνέπειες των μέτρων αυτών δυστυχώς έχουν μια δευτερεύουσα θέση. Ευχαριστώ κύριο Σαρόλα, 1,5 λεπτό. Επίτροπε, όταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε την φιλοδοξία του να πετύχει ένα τριπλό α για την Ευρωπαϊκή Ένωση, απέστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Θα πρέπει να δώσουμε εξίσου σημασία και στα κοινωνικά θέματα όσα αποδίδουμε και στα οικονομικά θέματα. Αυτή είναι ακριβώς η βάση μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς είναι ένας προσανατολισμός, είναι μια βούληση, πρέπει όμως να την κάνουμε πραγματικότητα. Τι δείκτες, τι παραμέτρους θα λάβουμε υπόψη μας για να αξιολογήσουμε τις πολιτικές και την πρόοδο. Προς την κατεύθυνση αυτή για να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε εφιώς να βασιστεί στους μηχανισμούς που υπάρχουν τώρα, όπως ε, οι μηχανισμοί Χέρις και Βιζεό στην Γαλλία ε, απαιτείται έτσι να υπάρξουν κάποιες σωστές ε, κατευθύνσεις αλλά αυτό δεν αρκεί όπως και για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις αποσπάσεις θα πρέπει να υπάρξουν υπηρεσίες επιθεώρησης ικανοποιητικές για να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν. Πρόκειται για μια ουσιαστική προσπάθεια για την αξιοπιστία της Ένωσης αλλά και για τη συμφιλίωση των πολιτών με την ευρωπαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ για ένα λεπτό η κυρία Τζεντήλε. Η πολιτική πρέπει να δίνει λογικές απαντήσεις στις φιλοδοξίες κοινωνικής ε, ισορροπίας. Από αυτό εξαρτάται η ποιότητα της ζωής των ανδρών, των γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ανέργων κάθε ηλικίας. Η φτώχεια προκαλείται από την έλλειψη πλούτου και θα πρέπει η Επιτροπή να δώσει γρήγορα απαντήσεις ξεπερνώντας αυτά τα οποία ζήσαμε μέχρι τώρα και αυτά τα οποία ακούσαμε σαν μια άχρηστη προπαγάνδα. Πρέπει να υπάρξει προώθηση των δικαιωμάτων, των ευκαιριών για τις πιο εύθραυστες κατηγορίες να λάβουμε μέτρα το ταχύτερο δυνατόν. Το θέμα δεν είναι μόνο να επηρεάσουμε και να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις αλλά τους πολίτες και ιδιαίτερα ακόμα και τους πολίτες αυτούς τους φτωχούς που χτυπούν την πόρτα μας και γι' αυτούς θέλουμε πολιτισμό, θέλουμε δημοκρατία, θέλουμε ειρήνη. Σας ευχαριστώ για 1,5 λεπτό η κυρία Σάντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Το 2014 ο πρόεδρος Γιούνκερ δήλωσε ότι θέλει να δώσει ένα τριπλό κοινωνικό άλφα στην Ευρώπη. Αυτή η δήλωση ήταν η απαρχή της συζήτησης και μετά από πάνω από ένα χρόνο πολλοί από εμά πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να δώσουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτου λεχθέντος παραμένει το θέμα του τι εννοούμε όταν λέμε κοινωνικό πρόσωπο. Κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη κοινωνική προστασία είναι το να έχει κανείς μια δουλειά, μια δουλειά αξιοπρεπή, μια δουλειά η οποία τον ανταμείβει σωστά. Αυτό απαιτεί να δώσουμε στους συμπολίτες μας όλα τα εργαλεία ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, δηλαδή να έχουν τις δεξιότητες, τις γλωσσικές δεξιότητες και την δυνατότητα να ακολουθήσουν την κινητικότητα της εποχής. Παράλληλα, θα πρέπει να δώσουμε τα ίδια εργαλεία σε όλους, χωρίς αθέμητο ανταγωνισμό, ε, χωρίς ε, να πλήττονται οι λιγότερο ισχυροί κοινωνικά. Εκ παραλλήλου θα πρέπει να επιτρέψουμε στις επιχειρήσεις, βιομηχανικές, γεωργικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις, να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Αυτό απαιτεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα είναι ευνοϊκό προς τις επιχειρήσεις, που θα τις ενθαρρύνει να επενδύουν και να καινοτομούν. Πίσω από το κοινωνικό τριπλό α, πίσω από το σλόγγαν του κοινωνικού αλφα θα πρέπει η Ευρώπη να μπορέσει μετά από την κρίση που συγκλώνησε τους πολίτες και που τους έβαλε σε μεγάλη επισφάλεια εργασίας, να γίνει η Ευρώπη μια Ευρώπη που θα συμφιλειωθεί εκ νέου με τις επιχειρήσεις και τους ε, υπαλλήλους, τους μισθωτούς και θα τίνει προς την κοινωνική σύγκληση. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό ο κύριος Μπαλάς. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε χρειαζόμαστε δείκτες στον οικονομικό τομέα και στον κοινωνικό τομέα για να μπορούμε να εξελιχθούμε. Θα ήθελα να σας πω την γνώμη μου επί του θέματος. Όταν έχουμε μια ελεύθερη εσωτερική αγορά, με ε, ε, ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, εάν παράλληλα δεν έχουμε και οικονομική και κοινωνική σύγκληση, απειλείται αυτή η εσωτερική αγορά. Και ακόμη πιο σοβαρό είναι το ότι αν δεν υπάρχει μια διαδικασία κοινωνικής σύγκλησης, τότε μπορεί να απειλείται και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η ε, εθνικιστικές φωνές κατά της Ευρώπης θα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη από ό,τι σήμερα. Γι' αυτό και απαιτείται μία μέθοδος, δηλαδή ότι πρέπει να προτείνετε κάποια θέματα, ακόμη και αν είστε μειοψηφία, ακόμη και αν το Συμβούλιο δεν συμφωνεί, εσείς θα πρέπει να προτείνετε θέματα στα οποία το, το Κοινοβούλιο θα σας, θα σας υποστηρίξει για να μπορέσουμε να κάνουμε πρόοδους. Και αν δεν μπορούμε και 28 να προχωρήσουμε, υπάρχει η Ευρωζώνη η οποία σιγά σιγά θα συμπαρασύρει και τους υπολείπους. Κυρία Τάισεν, λοιπόν, το κοινωνικό τριπλό Α δεν πρέπει να μείνει στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει μια μέθοδο. Ευχαριστώ. Ενάμιση λεπτό, κυρία Τόμς. είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα κοινωνικά θέματα παραμένουν σημαντικά στην ημερήσια διάταξη. Αυτό αυτός, στην Αυτός είναι ο λόγος στον οποίο μπορούμε να δούμε ότι η ιδέα αυτή του τριπλού κοινωνικού α περιλαμβάνει ό,τι μας, μας είναι σημαντικά. Εκπαίδευση, απασχόληση, καλύτερο συντονισμό των κοινωνικών συστημάτων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε μια πρωτοβουλία για ένα ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Η Ευρώπη ήταν και μένει μοντέλο κοινωνικών ε, δικαιωμάτων. Θα πρέπει να κρατά αυτό το, αυτή την πρωτοκαθεδρία ανά τον κόσμο. Για να γίνει ωστόσο αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το σύστημα αυτό και να έχουμε ένα σύστημα πιο αποδοτικό. Είμαι πεπισμένος ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα συμβάλλει σε αυτό. Πολλά ερωτήματα ωστόσο παραμένουν εκρεμή. Για παράδειγμα, πώς θα λειτουργήσει το σύστημα του τριπλού α. Αυτό είναι ο λόγος ε, που απευθύνομαι την ερώτηση αυτή στην ε, Επιτροπή. Περιμένω κύριε Επίτροπε την απάντησή σας. Για ένα λεπτό ο κύριο Τζανονάτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σημαντική η παρούσα συζήτηση για να διευκρινίσουμε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να περιοριστεί μόνο στην οικονομική διάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απορρίπτεται. Δεν μπορούμε να χτίσουμε μια κοινή αγορά χωρίς πολιτική και κοινωνική Ευρώπη. Πρέπει να υιοθετήσουμε δεσμευτικούς κοινωνικούς δείκτες σε συμφωνία με τα συνδικάτα βεβαίως και ενισχύοντας τον κοινωνικό διάλογο για να χτυπήσουμε το ντάμπινγκ επιβεβαιώνοντας ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να υπερισχύουν των οικονομικών ελευθεριών. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες βελτίωσης των συνδικών εργασίας και ζωής τους όπου και να ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό επίγει να ορίσουμε έναν σαφή μηχανισμό ελάχιστου εισοδήματο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνία με, τα, με τους κοινωνικούς εταίρους που έχει στόχο να περιοριστούν οι διαφορές αντιμετώπιση. Εγώ επίσης πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να δεσμευτεί το ταχύτερο δυνατό να εξετάσει τον αντίκτυπο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό. Ο κύριος Λαβρίγε, πρόεδρε, επίτροπε, συνάδελφοι. Τον Οκτώβριο του 2014 όταν μίλησε ο πρόεδρος και για το κοινωνικό τριπλό α έθεσε την Ευρώπη σε μια νέα δυναμική. Στον τομέα αυτό πρέπει να είναι παράδειγμα η Ευρώπη. Η κοινωνική Ευρώπη δεν πρέπει να μείνει μια ουτοπία. Βεβαίως ε, δεν μπορούμε να έχουμε ομοιόμορφο εργατικό κώδικα για 28 κράτη-μέλη, αλλά μπορούμε να έχουμε κοινά κριτήρια και σημεία αναφορά για όλου του εργαζόμενου. Αυτή η σύγκληση θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το κοινωνικό ντάμπινγκ και να απαντήσει στη δυσλειτουργία πολλών οδηγιών. Ξέρω ότι στο θέμα αυτό, Επίτροπε, έχετε ασχοληθεί σημαντικά με το θέμα της απόστασης των ε, τη απόσπαση εργαζομένων, αντικείμενο προηγούμενη συζήτηση, διορθώνοντα κάποιε ανεπάρκειε του υφιστάμενου κειμένου για να πετύχουμε την κοινωνική, την κοινωνική Ευρώπη πρέπει να ξεπεράσουμε τις δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να ξεκινήσουμε ένα κοινωνικό διάλογο όπως το είχε φανταστεί ο παλιός πρόεδρος της Επιτροπής Ζακ Στη Γαλλία η κοινωνική προστασία και τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν είναι κενά λόγια, αλλά δεν θα πρέπει να κάνουμε στην Ευρώπη όπως στη Γαλλία το λάθος να προσθέτουμε κανόνες. Οι επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να λειτουργούν και αποτελεσματικά. Επί της ουσίας ευχαριστώ. Κύριος Γκουτιέρες το ένα λεπτό. Πρόεδρε, πριν από 1,5 χρόνο ο Γιούνκερ μιλούσε εδώ για πρώτη φορά για το τριπλό κοινωνικό α. Και θυμάμαι γιατί είπε ότι το πρότεινε, για να αλλάξει η δυναμική ανάμεσα στην αντιμετώπιση των ε, πολιτών της ευρωπαϊκής πολιτικής ιδίως της περίοδου Μπαρόζο. Η έννοια της, ε, του τριπλού κοινωνικού α είναι για να δείξουμε ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όπου ο πολίτης ήταν στο κέντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ένα χρόνο μετά η, το, κοινωνικό, το τριπλό κοινωνικό α παραμένει ένας ε, όρος κενός περιεχομένου. Πρέπει να τον γεμίσουμε. Με, αυτό πρέπει να γίνει με τρεις τρόπους. Πρώτον, ε, ε, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ελάχιστων μισθών. Δεύτερον, ευρωπαϊκή ασφάλεια απασχόληση για να μοιραστεί αλληλεγγύη των ανέργων ανά την Ευρώπη. Και τρίτον, ελάχιστο εισόδημα ένταξη για να ξεριζωθεί ο κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτά είναι τρία βασικά δεδομένα για να γεμίσει περιεχόμενο το τριπλό κοινωνικό α και να κρατήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που ε, προστατεύει εκατομμύρια Ευρωπαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ενάμιση λεπτό η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ. Επίτροπε, άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον τις εξηγήσεις σας της έννοιας του τριπλού κοινωνικού αλφα αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δείχνει τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστασίας που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες πολιτικές αλλά και νέες πολιτικές και αναφερθήκατε σε αυτές. Να υπογραμμίσω εδώ την υποστήριξη την οποία θα πρέπει να δώσουμε στην προσπάθεια εξισορρόπησης της προσωπικής ζωής, της ατομικής ζωής και της σταδιοδρομίας οι νέες οικογένειες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να επενδύσουν στα παιδιά τους γιατί τα παιδιά τους είναι το μέλλον και η ευρωπαϊκή προοπτική. Πώς θα στηρίξουμε αυτούς τους νέους γονείς λοιπόν. Πώς θα στηρίξουμε αυτούς τους νέους ανθρώπους, αυτοί που ζητούν να υπάρξουν ε, ε, νέες μορφές προστασίας των εργαζομένων, να τους πούμε ότι απαιτούνται βέβαια και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και πετυχημένοι εργοδότες και αυτό θα δημιουργήσει ένα σταθερό νομικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου λοιπόν και εφόσον θέλετε να αναθεωρήσετε την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων θα πρέπει να το κάνετε αυτό προστατεύοντας το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο κύριος Σάιμον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για τον κοινωνικό πυλώνα της Ευρώπης ε, το περιέγραφε ε, ως ένα έγγραφο αναφοράς νομικού χαρακτήρα που εκφράζει τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν θα ισχύσει στα 9 από τα 28 κράτη-μέλη και αυτό φαίνεται κάπως περίεργο όταν μιλάμε για μεγάλες σημαντικές αρχές οι οποίες δεν θα ισχύσουν, δεν θα εφαρμοστούν σε εκατοντάδες εκατομμυρίων πολιτών. Θέλω να πω προς την Επίτροπο ότι ευτυχώς εσείς και ο Πρόεδρος Γιούνκερ δεν γράψατε το δευτερονόμιο, γιατί ε, αν είχατε γράψει τις δέκα εντολές ε, θα λέγατε ε, ου κλέψεις, ου φωνεύσεις και ου μοιχεύσεις, αλλά αυτό μπορεί να επιτρέπεται ή να είναι προαιρετικό στην Πολωνία αν είναι σημαντικές οι αρχές θα πρέπει να ισχύουν για όλους. Διαφορετικά δεν είναι παραλόγια για να κρατάτε τους σοσιαλιστές ευχαριστημένους χωρίς πραγματική ουσία. Οπότε ας μην σπαταλούμε το χρόνο μας. Αν όμως είναι αλήθεια αυτό το οποίο θέλετε να προτείνετε, κάπου στο έγγραφο θα πρέπει να αναφέρονται και οι θέσεις ποιότητας, οι ποιοτικές θέσεις εργασίας. Στην εκλογική μου περιφέρεια υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι με συνθήκες εκμετάλλευσης. Αυτό το έγγραφο θα πρέπει να αναφέρει και αυτούς τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. 1,5 λεπτό ο κύριος Βάντεν Κεντελάερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Είμαι νέος Ευρωβουλευτής και συντονιστής του ΕΛΚ και θα ήθελα να αναφερθώ στην κατάσταση των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενιαία αγορά και τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς για μένα θεωρούνται αυτονόητα. Έχουμε όμως τώρα την οικονομική και νομισματική κρίση και έχουμε κληρονομήσει μια δύσκολη κατάσταση. Η δική μου γενιά βλέπει ότι το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η Ευρώπη δεν προσδιορίζεται από την οικονομία αλλά από τον κοινωνικό χαρακτήρα. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιήσουμε τους νέους και αυτό απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Ένας στους πέντε νέους είναι άνεργος. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει το έναυσμα σε αυτή την πρωτοβουλία και υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία. Αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Το θεματολόγιο για τις νέες δεξιότητες, παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να εξεταστεί πολύ λεπτομερώς, όπως και η κινητικότητα. Χρειαζόμαστε μια κοινωνική Ευρώπη, όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν ίσα δικαιώματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πρέπει εμείς να είμαστε η γενιά που θα θυσιαστεί. Πρέπει να τονίσουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα και αυτό είναι καθήκον όλων μας. Ευχαριστώ πολύ και τώρα στη διαδικασία Catch the Eye έχω 7 ομιλητές, θα δώσω σε όλους το λόγο και ξεκινώ για ένα λεπτό, μην το υπερβείτε όμως, ένα λεπτό, η κυρία Γιασκαουέσκα, Ντανούτα Γιασκαουέσκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρο που μπορεί να μιλήσουμε για τρίπλο αλφα στην κοινωνική πολιτική σήμερα. Μας εξήγησε η Επίτροπος τι σημαίνει τρίπλο κοινωνικό αλφα και τι στόχους έχει. Ποιες, ποιες νομ, ποια νομοθετικά κείμενα θέλει να αλλάξει. Ωραία είναι αυτά. Αλλά δεν θα είναι εύκολο να το υλοποιήσουμε. Ξέρετε ότι η κοινωνική πολιτική επηρεάζει σοβαρά την ζωή των πολιτών και απαιτεί υπεύθυνη παρέμβαση και από τα κράτη και από την Ένωση. Ο στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη συνοχής στις κοινωνικές πολιτικές των κρατών μελών που θα επιτρέπουν αύξηση της καινοτομία, καλύτερη ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα εργασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφοροποιημένων αλλαγών στις πολιτικές των κρατών μελών. Ξέρουμε ποιες είναι οι προκλήσεις Θέλουμε να εισάγουμε νέα στοιχεία στην αγορά εργασίας. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ας δει η Επιτροπή δύο εκθέσεις που θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο, σημαντικές και δύο η αντιμετώπιση των στόχων της ε, φτώχειας, γνωμοδότηση και η φτώχεια από τη διάσταση της γυναίκας. Χρειαζόμαστε μεγάλη ορμή για να πετύχουμε τους στόχους κατά της φτώχειας με σημαντική κοινωνική έμφαση στο ευρωπαϊκό εξάμεινο με σαφή έμφυλη προοπτική. Είναι η μέρα της γυναίκας σήμερα. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσανάλογα μεγάλους κινδύνους αποκλεισμού και φτώχειας. Όταν αντιμετωπίζουμε την φτώχεια, ανεβάζουμε και τις γυναίκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δημιουργήσει μια κοινωνικά δίκαιη και ίση Ευρώπη, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες του φύλου για να πετύχουμε αυτή την, για να υλοποιήσουμε αυτά τα γεγονότα. Κύριος Μαριάς, ένα λεπτό κυρία πρόεδρε το τριπλό κοινωνικό α του κυρίου juncker έχει αποτύχει. έχουμε στρατιές ανέργων στην ευρώπη έχουμε φτώχεια στην ευρώπη έχουμε 9% ανεργία έχουμε μεγάλη ανεργία στους νέους έχουμε 25% ανεργία στην ελλάδα. αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια σωστή κοινωνική πολιτική χρειάζονται τρία τουλάχιστον πράγματα ευρωπαϊκό ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα ελάχιστος ευρωπαϊκός μισθός ευρωπαϊκό επίδομα ανεργίας. αντί να έχουμε αυτά έχουμε μια διαφορετική κατεύθυνση. όπως είπα προηγουμένως η τελευταία συμφωνία για την παραμονή της βρετανίας στην ουσία διαλύει κάθε κοινωνική πολιτική στην ευρώπη διότι δεν θα υπάρχει μόνο διακριτική μεταχείριση όσων ευρωπαίων εργάζονται στη βρετανία αλλά και όσων βρετανών θα εργάζονται στην ευρωπαϊκή ένωση διότι η κυρία μέρκελ είπε ότι της αρέσει αυτό το σύστημα. επομένως δεν έχουν εξηγηθεί καν στους βρετανούς πολίτες ότι όταν αυτοί θα είναι εργαζόμενοι στην ευρώπη θα μπορούν να γίνεται διακριτική μεταχείριση εις βάρος τους. Thank η... στην ουσία η προσπάθεια την οποία έκανε ο κύριος Γιούνκερ για το κοινωνικό τριπλό α ε, δεν είναι κάτι το οποίο έχει ουσιαστική σημασία. Ταυτόχρονα αυτό το οποίο επιδιώκει η πολιτική αυτή είναι η λιτότητα. Ε, ξέρουμε ότι δεν βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας, ίσα ίσα μη ε, χειροτερεύουν και ξέρουμε επίσης τι γίνεται και στην περίπτωση της ανεργίας των νέων. Το τριπλό κοινωνικό α λοιπόν είναι κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να οδηγήσει σε μέτρα περισσότερο υπέρ του κεφαλαίου και όχι υπέρ των πολιτών, κάτι το οποίο θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την ανεργία θα πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης με συγκεκριμένα δικαιώματα γιατί αλλιώς θα οδηγηθούμε στην θανάτωση των κοινωνικών μας συστημάτων. Ο κύριος Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τον Οκτώβριο του 2014 Άκουσα με μεγάλη ικανοποίηση τη δήλωση του κυρίου Γιούνκερ με την ιδέα του κοινωνικού τρίπλου Α. Είμαι υπέρ της αρμονικής οικονομικής ανάπτυξης που απαιτεί παράλληλα και δράσεις για τη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης και της απασχόλησης των πολιτών. Η κοινωνική βαθμολογία θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ένας γενικός στόχος ή έκφραση γενικών απόψεων. Χρειαζόμαστε και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να επιτύχουμε το τριπλό α. Καταρχήν χρειαζόμαστε δείκτες που θα είναι εύκολα μετρήσιμοι για να παρακολουθούμε την πρόοδο και ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα υποβάλει σχετικές προτάσεις. Σημειώστε επίσης ότι οι δράσεις για το κοινωνικό τριπλό Α θα πρέπει να απευθύνονται εξ αρχής σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο σε μέρος αυτής. Ο επόμενος ομιλητής, χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή μιλάει για τον αθέμητο και ελεύθερο ανταγωνισμό και θεωρεί ότι αυτό αποτελεί τη βάση της κοινωνικής πρόοδου. Σήμερα στην Ευρώπη ο ανταγωνισμός νομίζω δεν είναι ούτε ελεύθερος ούτε αθέμητος, διότι τα κοινωνικά συστήματα είναι εξαιρετικά διαφορετικά μεταξύ των διαφόρων χωρών. Η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες για την κοινωνική Ευρώπη και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε. Με την γεωργική κρίση, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι δημιουργούνται στρεβλώσεις ανταγωνισμού με τη χρήση των αποσπασμένων, όπως αποκαλούνται αυτοί οι εργαζόμενοι, και αυτό οξύνει την κρίση στην γεωργία. Θεωρώ ότι πρέπει να εναρμονίσουμε την Ευρώπη σήμερα, με, να εναρμονίσουμε την κοινωνική νομοθεσία. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι θα πρέπει και το φορολογικό δίκαιο να εναρμονίσουμε, γιατί αυτά είναι τα προβλήματα της Ευρώπης. Έλλειψη της κοινωνικής εναρμόνισης και της φορολογικής εναρμόνισης. Ευχαριστώ, κ. Πόλτσακ. Ευχαριστώ. Για άλλο θα μιλούσα. Ο προηγούμενος ομιλητής ωστόσο μου άλλαξε τον λόγο. Νομίζω ότι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα δημιουργήσει αύξηση της κοινωνικής προστασίας. Η... Μια οικονομικά ισχυρή Ευρώπη δεν σημαίνει ότι θα μπορέσει να παράσχει κοινωνική προστασία. Σε ό,τι αφορά τα μέσα που έχουν τα κράτη-μέλη στην διάθεσή τους, αντίθετα από τον προηγούμενο μιλητή, πιστεύω πως είναι σημαντικό να παρέχουμε στα κράτη-μέλη κάποια δυνατότητα διαφυγής. Δεν μπορούμε να νομοθετούμε τελείως δεσμευτικά και να μην αφήνουμε κάποιες ευκαιρίες ευελιξίας στα κράτη-μέλη. Η Επίτροπος έχει το λόγο. Eh, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω για τον πλούτο των παρεμβάσεων. Σας άκουσα πολλές παρατηρήσεις, υποστηρίζετε την ιδέα του τριπλού κοινωνικού α. Διαπιστώνω επίσης ότι επιθυμείτε να λάβουμε πιο συγκεκριμένες αποφάσεις για το τι χρειάζεται. Και αυτή την προσπάθεια την έχουμε ξεκινήσει. Βέβαια προβλήματα έχουμε, τα οποία δεν περιμέναμε να είμαι ειλικρινής συμφωνείτε με τις ανησυχίες που έχω σχετικά με τις συνέπειες της κρίσης. Υπάρχει μια αύξηση της φτώχειας, ενώ στόχος ήταν η μείωση. Είδαμε όμως να αυξάνεται. Ευτυχώς μειώνεται η ανεργία των νέων μήνα με μήνα. Πάντως πολλά μένει να γίνουν, γιατί είναι ακόμα πολλοί οι άνεργοι νέοι και έχουμε επίσης προβλήματα με τη μακροπρόθεσμη ανεργία. Όσο πιο διασπασμένη είναι η αγορά εργασίας, τόσο χειρότερη και ανεξέλεγκτη γίνεται η κατάσταση. Είναι σαφές λοιπόν ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Πρέπει να κατανοήσουμε ποιες είναι οι προκλήσεις. Υπήρξε μια κρίση, αλλά από τότε δεν σταμάτησε να γυρνάει ο κόσμος. Υπάρχουν περαιτέρω προκλήσεις, η οικονομία αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, υπάρχουν προβλήματα δημογραφικά, αλλαγές σε επίπεδο οικογενειακής διάρθρωσης, υπάρχει ψηφιοποίηση, παγκοσμιοποίηση, νέοι τρόποι απασχόλησης, τα νέα business model, δεν είμαστε εναντίον όλων αυτών, αλλά θα είμαστε ε, σωστοί, ενήμεροι, έτσι ώστε η κοινωνική πολιτική να βοηθήσει αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη από προστασία περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Οι απαντήσεις μας θα πρέπει να έχουν σαν στόχο να επανέλθουν οι άνθρωποι αυτοί στην αγορά εργασίας. Απαιτείται περισσότερη σύγκληση, γιατί όσο περισσότερες ανισότητες υπάρχουν αυτό δημιουργεί προβλήματα στην οικονομική ανάπτυξη, μειώνει τις προοπτικές και αυτό είναι ο βασικός μας στόχος. Είναι δύσκολο να δώσουμε βέβαια τη σωστή απάντηση. Υπάρχουν επίσης τα θέματα της ισότητας ευκαιριών, της ισότητας στην πρόσβαση εργασίας, Υπάρχει το θέμα των ικανοτήτων, δεν είναι μόνο θέμα μαθητείας ε, κατά τη διάρκεια της ζωής, αλλά υπάρχει και το θέμα της δυνατότητας αλλαγής ε, γνώσεων ικανοτήτων. Και υπάρχει θέμα επίσης και με την βελτίωση της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής ασφάλισης. Το θέμα δεν είναι να είναι βιώσιμα τα συστήματα, αλλά να είναι αποτελεσματικά να καταπολεμούν τους κινδύνους, να καλύπτουν πραγματικά και να επιβάλλουμε, θα έλεγα, ικανοποιητικές συνθήκες απασχόλησης. Σε αυτά δεν μπορούμε να απαντήσουμε μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει από κοινού να έχουμε ένα κοινό όραμα για να υπάρξει μια κοινή απάντηση. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο ε, μέσω ανάληψης της ευθύνης από την πολιτική. Αυτό γίνεται. Απαιτείται όμως να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Οι κοινωνικοί εταίροι είναι αυτοί που θα μας επιτρέψουν να βρούμε τις καλύτερες λύσεις και θα μας επιτρέψουν να τις εφαρμόσουμε με σωστό τρόπο. Η προσπάθεια θα πρέπει να γίνει από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους πολιτικούς υπευθύνους και θα πρέπει όλοι μαζί να εξετάσουμε το πακέτο αυτό που ξεκίνησε σήμερα, να υπάρξει μια προσεκτική ανάγνωση, εξηγούν τι είναι ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Διαβάστε τα παρακαλώ, διαβάστε και τα παραρτήματα για να καταλάβετε σε τι ε, θα μοιάζει ο πυλώνας αυτής. Υπάρχουν επίσης και δύο κείμενα εργασίας, δύο staff working documents που αναφερόμαστε στο πρωτογενές δίκαιο, στο διεθνές δίκαιο, στο μη υποχρεωτικό δίκαιο, δεσμευτικό δίκαιο. Ε, είναι μια σειρά από στοιχεία στα οποία γίνονται συγκεκριμένες αναφορές τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεχθούν τις προτάσεις αυτές και να τις εφαρμόσουν και να δούμε επίσης και τι γίνεται με τις οικονομικές τάσεις και προοπτικές. Σας ευχαριστώ λοιπόν, μελετήστε τα παρακαλώ, ζήτησα και από τα κοινοβούλια, τα εθνικά και από τις κυβερνήσεις και από την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή να συνεισφέρουν στην επεξεργασία της προτάσεως αυτής για να καταλήψουμε σε ένα έγγραφο το οποίο θα διασφαλίσει την κοινωνική ειρήνη και την κοινωνική Ευρώπη. Η κοινωνική Ευρώπη, όπως είπε ο κύριος Βανκάντελάρε, θα είναι μια Ευρώπη που θα δώσει τη δυνατότητα να ζήσουν με σωστό τρόπο τα παιδιά της. Έτσι θα προχωρήσουμε στην οικονομία, την κοινωνική της αγοράς. Αν πετύχουμε το 3α θα το αξίζουμε και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα. Η οικονομική ανάπτυξη είναι απαραίτητη. Πρέπει να καταστεί εφικτή και να εφαρμοστεί. Αλλά θα πρέπει να οδηγεί στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και στη σωστή προστασία των εργαζομένων. Δεν πρέπει να παίζουμε με τις λέξεις, δεν πρέπει να αερολογούμε, πρέπει όμως να αναλάβει ο καθένας τις υποχρεώσεις του και τότε μόνο θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με σωστό τρόπο. Ο πυλώνας λοιπόν αυτός ο κοινωνικός που ξεκινάει σήμερα νομίζω ότι είναι μια σωστή πρόταση. Αυτοί οι οποίοι μας λέγουν ότι η κοινωνική Ευρώπη δεν υπάρχει, ότι έχει χάσει το ραντεβού με την ιστορία, δεν είναι σωστό. Εγώ ήμουνα ευρωβουλευτής, έχω εργαστεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν υπάρξει προπαρασκευαστικές εργασίες πριν ξεκινήσει η προσπάθεια για την κοινωνική Ευρώπη του μέλλοντος. Ας ανασηκώσουμε τα μανίκια μας λοιπόν και ας εργαστούμε και τότε μόνο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα και έτσι αυτοί που έρχονται εδώ θα βρουν μια Ευρώπη όπου αξίζει κανείς να ζει με ισότητα ευκαιριών και αυτοί που έχουν κάποια προβλήματα, έχουν λιγότερες ικανότητες ή έχουν κάνει λάθη στο παρελθόν θα μπορούν να παραμείνουν ανάμεσά μας μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος κοινωνικής προστασίας. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή και ελπίζω να συνεχίσουμε την συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Αποφασιστική η τοποθέτησή σας. Αλλάζουμε τώρα. Η Επίτροπος Γιώργο θα έρθει για την επόμενη έκθεση. Είναι όλοι εδώ. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση γιατί τώρα θα εξετάσουμε την έκθεση κινητή της ε,